non arriva il ministro Kunders. Και ήρθε ο υπουργό, ο κ. Κούντερ. Sì, buonasera. Allora, la... Καλησπέρα σας, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα σύμφωνα με την μελισσία διάταξη έχουμε τις δηλώσεις της αντιπροσώπου, της αντιπρόεδρου της Επιτροπής, υπάρτης εκπροσώπου για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια όσον αφορά την κατάσταση στο Μπαγκλαντέ. Και ευθύ αμέσω δώσουμε το λόγο εις, τον εκπρόσωπο της ε, Αντιπροέδρου. Τον λόγο έχει ο κύριος Κούντερς. Καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Πρέπει Ο Υπουργό χωρί μικρόφωνο. Και ο πρόεδρο χωρί ε, μικρόφωνο. Α, πέστε μου, πέστε μου πώ γίνεται, γιατί δεν το ξέρω. Α το ανάψει κάποιο άλλο το μικρόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μπαγκλαντές από πολύ καιρό είναι εταίροι και η σχέση μας οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι αμοιβαίο ωφέλιμα ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη αλλά και το εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος προορισμός, ο βασικός για τις αγωγές της χώρας και έχουμε πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις στην ε, χώρα και έχουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουμε και όλα αυτά συνέβαλαν στην ανάπτυξη για την χώρα και για κάποια επιτεύγματα όσον αφορά την ε, φτώχεια και την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Η σχέση μας με τη χώρα συνεχώς εξελίσσεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Μπαγκλαντές εντοπίζουν τις νέες προκλήσεις και έτσι ε, έχουμε την ανάπτυξη της ε, βιομηχανίας της τη ε, της χώρας. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια έχουμε τον πρώτο διάλογο με τη χώρα για την ε, διαχείριση της μετανάστευσης ε, στις 5 Απριλίου του 2016 και έχουμε σημαντικούς στόχους πολιτικής μας για το Βαγκλαντές. Μέχρι το 2021 η χώρα θα έχει βγει από τη φτώχεια, θα γίνει μια χώρα μέσου εισοδήματο. Να, ο βασικό στόχο που θα επιτευχθεί, φιλόδοξος ο στόχος, αλλά χρειάζεται να είναι όλοι αποφασισμένοι, όλοι να εμπλακούν στη χώρα, όλα τα θεσμικά όργανα και όλοι οι εταίροι τη χώρα διεθνώ. Έχουμε τώρα κάποιου είδου ανισχυτικέ όμω πολιτικέ εξελίξει που μπορεί να καταστρέψουν τι προσπάθειε και είχαμε αυτές τις ε, πίμεξους του 14, τις μποϊκοτάρες, η αντιπολίτευση, τις επέκρινε η διεθνής κοινότητα, οπότε τα πολιτικά, τα πολιτικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά τώρα είναι σε μια κατάσταση επιδεινούμενη, οπότε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Μαγκλαντές τελευταίας ε, διετίας, κάλυψε και τις εκλογές, αυτές που είπαμε, κάλυψε την καταστολή της ελεύθερης έφρασης των δικαιωμάτων και η Πάτη εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, οι ε, <clears throat> εκπρόσωποι της έχουν επισημάνει και κατακρίνει το ότι υπάρχει ακόμη θανατική ποινή και ε, επίσης δολοφονούνται ακτιβιστές και διάφοροι ε, ανεξάρτητοι παράγοντες αντιπολίτευσης οπότε βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξανόμενο προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί μια συνένεση, να οικοδομηθεί στη χώρα υπέρ δημοκρατίας, δικαιωμάτων, ελευθερίας έκφρασης, ελευθεριών και όλα αυτά να αποκατασταθούν στη χώρα και θα πρέπει να σταματήσει η αυθαιρεσία, η σύλληψη αντιπολιτευομένων, να υπάρξει ανοχή και επίσης ο χώρος και το βήμα για δημόσια συζήτηση. Η ελευθερία έκφραση είναι θεμελιώδες δικαίωμα αυτό. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των πολιτών να σταματήσουν ε, κάποιους αποτρόπες ε, επιθέσεις και ανθρωποκτονίες των πολιτών. Θα πρέπει επομένως οι ένοχοι να προσαχθούν στην δικαιοσύνη. Ήρθε η ώρα η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές όπως και τα δημοκρατικά κόμματα να συνοηθούν, να δεσμευθούν για έναν αυθεντικό διάλογο όσον αφορά τη σταθερότητα της χώρας και την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας. Χρειαζόμαστε ένα Μπαγκλαντές όπου όμως να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα οικονομικά δικαιώματα. Όλα αυτά θα πρέπει να προστατευτούν, αλλά θα πρέπει οι θεσμικοί όργανοι της χώρας να σέβονται το κράτος δικαίου, να εξασφαλίζουν προστασία για όλο τον πληθυσμό της χώρας. Άρα η ανοχή, η ανεκτικότητα, η ελευθερία θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Βεβαίω η κυβέρνηση της χώρας έχει να διδερματίσει σημαντικό ρόλο και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και Επίσης θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την κυβέρνηση. Υπολογίζουμε στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές μας τις προσπάθειες, Πρόεδρε. Με ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τώρα θα τοποθετηθούν οι πολιτικές ομάδες. Πρώτος ο κύριος Πρέντα για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για, συμμετέχω στην Επιτροπή για τον Μπαγκλαντέ και ανησυχώ για τι ανθρωποκτονίε και τη βία που ισχύουν στον Μπαγκλαντέ τελευταία. όπω γνωρίζετε, στον Μπαγκλαντέ υπάρχουν πολύ σκεφτικές μειονότητες, χριστιανοί, σούφοι, βουδιστέ κλπ. Υπάρχουν όμω και εκείνοι που είναι υπέρ ε, του πλουραλισμού του θρησκευτικού και του κοσμικού κράτου. Κάποιοι από αυτού δολοφονούνται, δέχονται επιθέσει, απειλούνται. Εκείνοι που υπερισπίζονται, παραδείγματο χάρη, την ελευθερία τη έκφραση, βλέπουν να απειλείται η ζωή του από ριζοσπάστε, από εξτρεμιστέ. Το κοινοβούλιο μα απέφθινε έκκληση το Νοέμβριο του 2015 από τι αρχέ του Μπαγκλαντέ επ' αυτού να γίνουν έρευνε ανεξάρτητε όσον αφορά αυτά τα εγκλήματα που διαπράσσονται. Να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά ε, τον εντοπισμό και την δίωξη των ενόχων. Οι αρχέ του Μπαγκλαντέ μα είπαν ότι θα έχουν μηδενική ανοχή έναντι των φρικαλαιοτήτων αυτών που διαπράττονται και να, ότι θα επικρατήσει ασφάλεια για τι μειονότητε. Ξεκίνησαν και έρευνε για κάποιε υποθέσει Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν περιμένουμε αποτελέσματα. Όπω έλεγε και ο υπουργό, αληθεύει ότι στο Μπαγκλαντέ η κατάσταση είναι όλος ιδιαίτερη από πλευρά πολιτική. Στις τελευταίες εκλογές ε, έγινε μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση και ε, αυτό ε, αυξάνει περισσότερο τις εσωτερικές συγκρούσεις. Πρέπει να ακυρώθηκε η αποστολή για τις εκλογές των Μπαγκλατές. Ε, ε, είχαμε αυτό το μποϊκοτάρισμα των εκλογών και αυξήθηκαν τελικά λόγω αυτών οι εντάσεις. Όλοι έχουμε επίγνωση της σημασίας του Μπαγκλαντές. Είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε από τους εταίρους μας όμως να βελτιωθεί σημαντικά το πολιτικό κλίμα και γενικά το κλίμα που επικρατεί στο Μπαγκλαντές. Λοιπόν, εν ονόματι των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γκίλ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον 10 ακτιβιστές δολοφονήθηκαν στον Μπαγκλαντές από τις αρχές του 2016. Το Ντάες και η αλ έχουν κάνει πολλές επιθέσεις. Όμως οι αρχές του κράτου συστηματικά αρνούνται να δεχθούν την παρουσία αυτών επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις φρικαλαιότητες για εκλογικούς σκοπούς αντί να προστατεύουν τους ακτιβιστές και βάλωτες ομάδες όπως είναι η ΛΟΑΔ. Έχει αποτύχει το Δικαστήριο του Διεθνέ των Εγκλημάτων του Μπαγκλαντές να εξηχνιάσει υποθέσεις. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Μπαγκλαντές να καταρρεύσει εντός των βιωτήτων. Πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα. Η Ινδία θα μας βοηθήσει. Έτσι θα σταματήσουμε να γίνει ακυβέρνητη η χώρα και να επικρατήσει η τρομοκρατία εκεί. Θα πρέπει όλα τα μέσα στον Μπαγκλαντές, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα τα σημερινά και αυτά που έγινε το 1972. Έξω δικαστικές δολοφονίες και συλλήψεις αυθαίρετες να σταματήσουν. Η ύπατη εκπρόσωπος πρέπει να ηγηθεί στον ΟΗΕ, να γίνουν και άλλα βήματα, να επιβληθούν κυρώσεις προς υπευθύνους για τις καταχρηστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις πλευρές. Πρέπει να υπάρχει δικαστικός διεθνής μηχανισμός που θα εξασφαλίσει το ότι θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη. Ο κύριος Τάνοκ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο, κύριε Πρόεδρε, το Μπαγκλαντές είναι κοσμικό κράτος δημοκρατίας νοτελικής Ασίας, είναι πολιτικό μοντέλο που υποστηρίζω. Ε, έχει θρησκευτική ανοχή, προστατεύει την ελευθερία τη έκφραση, τα δικαιώματα των γυναικών, την παιδεία, είναι αξίε που θα αναγνωρίζαμε και θα ε, τιμούσαμε στην Ευρώπη. όμω αυτέ οι αξίε απειλούνται στον Μπαγκλαντές σε αυτή τη φάση, αλλά όχι από την κυβέρνηση όπω κάποιοι διατείνονται εδώ σε αυτή την αίθουσα, αλλά από Ισλαμιστέ εξτρεμιστέ. Το 1971 η Τζαμάτα Ισλαμή σωστά απαγορεύτηκε στον Μπαγκλαντές, όχι μόνο οι Ισφρικαλαιότητε που διαπράχθησαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, αλλά και λόγω συνεχού ιδεολογική εκστατεία και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κατά του κοσμικού κράτου. Μετά την άσυλη απαγορεύσεω το 1979, η Τζαμάρ εξακολουθεί να ακολουθεί αυτό το μονοπάτι και έχει και σχέσει με τζιχατιστικέ ομάδε άλλε. Και παροτρύνω σήμερα το κόμμα στην πολίτηση, το BNP, να, στα... να καταγγείλει σχέσεις μαζί τους, ούτω ώστε να μπορέσει να παίξει το δημοκρατικό του ρόλο στην αντιπολίτευση. Μόλι το πρωί το, ένας ιερέας Ινδού ε, βρέθηκε νεκρό κοντά στο ναό. Η δολοφονία έγινε λόγω τη σχέση του και πολλοί άλλοι έχουν δολοφονηθεί σε παρόμοιε περιπτώσει, πανεπιστημιακοί, ακτιβιστέ, προστάτε των δικαιωμάτων των γκέι, bloggers ε, και άλλα, χριστιανοί, βουδιστέ, ε, και άλλοι εκπρόσωποι μειονότητων συστικών. Είναι από τι χώρε χώρες στον κόσμο το Μπαγκλαντέ και δεν απολαμβάνει τις πολυτέλειες ε, σωστά εκπαιδευμένη αστυνομία και υπηρεσιών ασφαλεία όπω εδώ στη Δύση. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολεμάμε κατά των δικών μα εξτρεμιστών και έτσι θα πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη και συμπάθεια προ την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ και λιγότερες επικρίσεις και καταδίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Σάκε. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Αγαπητή Πρόεδρε, Υπουργέ Κούρνερς, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να, να καταγγείλω σήμερα τις βαρύτατες ε, παραβιάσει των δικαιωμάτων, ε, τα αθώα θύματα που θρυνούμε. Δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη απάντηση. Έχουμε να κάνουμε με όλο και εντυνόμενα φαινόμενα. Εχθές μόλις ένας ενδουιστής ε, ιερέας σφαγιά κατακριουργήθηκε. είναι σαφείς οι ενδείξεις πως πίσω από αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα κρύβονται ακραίοι τρομοκράτες, Ισλαμιστές. Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει άλλη αιματοχυσία. Και μπορεί να βλέπουμε κάποιες δράσεις κατά τρομοκρατικών ομάδων, αλλά πολλά ακόμα θα μπορούσαν να γίνουν. Και όπως και να έχει, οι εκτελέσεις υπόπτων δεν είναι τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος που έχουν ε, των θυμάτων των Ισλαμιστικών ε, ομάδων, ένοπλων ομάδων ε, για μήνες τώρα και φοβούμε ότι δεν έχουμε αντιδράσει όπως θα έπρεπε. Πολύ σωστά επισημάνατε τους σημαντικούς δεσμούς, το εμπόριο, την ανάπτυξη, έχουμε και αυτά σταθμίσει στο παρελθόν. Όταν είχαμε τις καταρρεύσεις ε, των κτηρίων ε, εργοστασίων, ασκήσαμε την πίεση που μας επιτρέπει το δικό μας βάρος. Και τώρα λοιπόν πρέπει να το πράξουμε αυτό. Γιατί, γιατί κύριε Υπουργέ δεν μας ενημερώνετε περισσότερο, γιατί δεν μας λέτε ε, τι βήματα έχει αναλάβει ε, η είπατε εκπρόσωπος Μογκερίνη σε σχέση με τις αρχές του παγκλοντές και τι είδους συνέπειες μπορεί να υπάρξουν έχετε υπολογίσει εάν τυχόν δεν αντιδράσουμε επαρκώς σε αυτούς τους απετρόπιους φόνους τι γίνεται σε σχέση με το προσωπικό μας εκεί στις υπηρεσίες Ευχαριστώ Σάντσες Καλντελ ένα λεπτό Ευχαριστώ Πρόεδρε η Υπουργέ μετά από την ε, τραγωδία της Ράνα Πλάσα είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ασφάλεια εκεί σε αυτούς τους χώρους και είπαμε ότι έχουμε πάνω από χίλιους που ήταν σε αυτό το εργοστάσιο που υπηρετούν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες οπότε θέλουμε να τηρηθούν κάποιες δεσμεύσεις. εξαρτώνται τώρα από την καλή θέληση των ε, εταιριών. Δηλαδή τι βάλαμε την Αλεπού να φυλάξει τα κοτόπουλα η Μπένετον ή άλλες εταιρείε αρνούνται να δώσουν αποζημίωση στα θύματα εκείνης της τραγωδίας. Θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Κατεπηγόντως χρειάζεται νομοθεσία δεσμευτική και να υπάρξουν συνέπειες και στην πολιτική και στην ποινική δικαιοσύνη να τηρηθούν τα όσα προβλέπονται από τον ΟΗΕ. Πρόκειται να συνεχιστεί η διαδικασία και θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε και να μην είμαστε φραγμός γιατί έχουμε μεγάλη ευθύνη για το όσο γίνεται στο Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ Λάμπερτ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πρέπει να πω ότι ομιλώ ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με χώρες της Νότιας Ασίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Μπαγκλαντές. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, συντριπτική, η συντριπτική πλειονότητα των ε, Μπαγκλαντεσιανών ε, αισθάνεται η περηφάνεια που είναι τόσοι οι πολυμορφία στην κοινωνία τους και ανησυχεί ιδιαίτερα για την όξυνση και την κλιμάκωση ε, της κατάστασης από εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι Ισλαμιστές ή ότι ε, αποτελούν παρακλάδια της Αλκάιδα. Ε, είδαμε φόνους φρικτούς και επιθέσεις κατά ε, ΛΟΑΔΜ όπως επίσης και πιο πρόσφατα τον φόνο της συζύγου ενό αστυνομικού της αντιτρομοκρατικής. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δηλώσεις 100.000 ε, κληρικών με, τη, με τον ΦΕΤΦΑ για την ειρήνη που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε μερικές μέρες. Ε, προς αυτούς πρέπει να στραφούμε, πρέπει να καλλιεργήσουμε την ειρήνη, τις βάσεις της ειρήνης και όχι τις βάσεις του προβλήματος. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το έργο εκείνων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια την ελευθερία γιατί πολλοί δημοσιογράφοι μπαίνουν στη φυλακή αυτήν την εποχή. Χρειάζεται επίσης αποτελεσματική αστυνόμευση, σύστημα δικαιοδοτικό ε, ώστε να, να εξασφαλίζεται η ισότητα των πολιτών αντί του νόμου. Είναι για πολλούς ενισχυτική η κατάσταση και πρέπει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση στις προσπάθειές της. Μεν, ταυτόχρονα όμως καλώντας την να υπηρετήσει το συμφέρον όλων των Μπαγκλαδεσιανών. Ευχαριστώ πολύ. καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κλιμάκωση στον Μπαγκλαντές, άκρως ανησυχητική. Και διρωτάτε κανείς γιατί. Γιατί μια χώρα που διακρινόταν πάντα από την ανοχή, από την συγκατημένη θέση της πλειοψηφία των μουσουλμάνων έχει αυτή τη κατάσταση τώρα. Κυρίως οφείλεται στη φτώχεια. Ξέρουμε πόσο οι πολυεθνικές οι ευρωπαϊκές εκμεταλλεύονται κυρίως το ρύζι, τη γεωργία και τα εφαντουργικά και τους, για την εφαντουργία του εργαζομένου των Μπαγκλαντές και αυτό είναι κάτι που διευκολύνει τη δουλειά του Ντάις και της Αλκάιντα, τις εξτρεμιστικές αυτές ομάδες που δυσδύουν όλο και περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών εκεί στον Παγκλαντές. και οδηγούνται στη ριζοσπαστικοποίηση. Σαν Ευρώπη πρέπει να προωθήσουμε μεταρρυθμίσει στο δικαστικό τομέα. Καλύτερη λειτουργία τη αστυνομία. Πρέπει να ζητήσουμε πρόοδο όσον αφορά την δημοκρατία και την ελευθεροτυπία. Πρώτα να κάνουν λογαριασμού όμω με τι δικέ μα δράσει. Η οικονομική και κοινωνική σταθερότητα τη χώρα είναι βασικό πυλώνα για να εμποδιστεί η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση. Μην το λησμονούμε. Χρειαζόμαστε συνεκτική χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν συνεκτικέ πράξει και κινήσει από πλευρά των πολυεθνικών. Συνάδελφε Ρούε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Όπω γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, εδώ και τρία χρόνια το εργοστάσιο στη Ράνα Πλάζα κατέρευσε και 1.100 άνθρωποι ε, σκοτώθηκαν και 2.500 τραυματίστηκαν. Είναι μεγαλύτερο εγωγέα ε, βαμβακιού το Μπαγκλαντέ και το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών πάει στην Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν την καταστροφή ότι χρειάζεται συγκεκριμένη ε, δράση για να βελτιωθεί η ασφάλεια των κτηρίων και οι συνθήκε εργασία για του εργαζομένου. Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα αλλά και σε άλλε χώρε που προμηθεύουν ε, με προϊόντα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δύο χρόνια μετά από την υπογραφή του Συμφώνου Σταθερότητα, είδαμε πολύ θετικέ υποχρεώσει που ανέλαβε η κυβέρνηση τη χώρα, του Μπαγκλαντέ. Όμως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση κυβέρνηση να σέβεται τη Σύμβαση 87 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και να καλύπτεται νομικά, να καλύπτονται και ελεύθερες ζώνες, οι εξαγωγικές ζώνες και θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Χρειάζεται σωστός έλεγχος των χώρων εργασίας και να πληρούνται οι προδιαγραφές του ILO. Ελπίζω ότι αυτό το σύμφωνο τελικά θα έχει θετική ε, επίδραση στην κατάσταση. Και αυτή η χώρα θα πρέπει να είναι παράδειγμα για άλλες ε, χώρες και ελπίζω ότι θα, η διεθνής κοινότητα θα κινηθεί πιο συντονισμένα στο μέλλον. Έχετε το λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση στο Παγκλαντές και ο κίνδυνος εμφυλίου δεν αποκλείεται. Χρόνια τώρα είναι δύο, με, δύο μέτωπα, το ένα απέναντι στο άλλο. Συνεχίζεται και κλιμακώνεται η βία και βέβαια οι εξτρεμιστές αξιοποιούν την κατάσταση αυτή. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οργανώσεις όπως οι χαότικα έχουν ε, βρεθεί σε κίνδυνο ακόμη και εξαφάνισης, έχουμε την κατακρεούργηση ενός ενδουιστή αερέα, ιερέα και πολλά άλλα τέτοια κλίματα. Είναι δυνατόν ακόμη να σταματήσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο της βίας. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ η Ευρώπη. Γιατί η φωνή της Ευρώπης ακούγεται στο Μπαγκλαντές. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ντέμες Μάκερ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, όντω ε, είναι βάσιμη η φόβη και ανησυχίε για το Μπαγκλαντέ. Είναι όλο και πιο κατασταλτική η δράση των αρχών ε, κατά των μέσων μαζικής ενημέρωση, των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ένα φονταμενταλιστικό κίνημα του Ισλάμ προσπαθεί να ρίξει ρίζες στο Μπαγκλαντές και φαίνεται ότι δεν γίνονται αρκετά για να σταματήσουν αυτές οι αστρεμιστικές τάσεις. Εάν συνεχίσει λοιπόν το Μπαγκλαντές να παρασύρεται προς την ακρότητα αυτή θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις και συνέπειες. Ιδιαίτερα θέλω να συμφωνήσω με την έμφαση την οποία δίνεται στο ότι είμαστε πολύ σημαντικός εταίρος, κύριος εμπορικός εταίρος και ο μεγαλύτερος αγοραστής των ε, προϊόντων της υφαντουργίας του Μπαγκλαντές και το Μπαγκλαντές έχει το δικαίωμα να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τελωνιακούς δασμούς. Είναι κομμάτι της συμφωνίας τα πάντα ε, πλήν των όπλων και νομίζω ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν πράγματα εκεί όπως είδαμε με την περίπτωση του Ράνα Πλάζα. Μπορούμε να πιέσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε και για τη σταθεροποίηση, την κοινωνική συνοχή και ε, την εξομάλυνση. Ο κύριος Τόμας Μάν, ευχαριστώ. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Μπαγκλαντές είναι πολύ ενισχυτική. Η πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται από διαρκή αντιπαράθεση των Ερβάρμι Πιλίκ και του BNP. Βλέπουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ Σαν Καζίνα και Καλεντατσία και έχουμε και πολλούς φόνους από ακραίους φανατικούς έναν βίο πόλεμο κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, των blogger, των αλλοδαπών. Ένα σύστημα δικαιωματικό το οποίο έχει τόσο πολύ κομματικοποιηθεί που δεν μπορεί να λάβει σωστές αποφάσεις, που όλο λαμβάνει εισφαλμένες αποφάσεις. Το κράτος δικαίου λοιπόν, ο δημόσιος διάλογος, η ελευθερία της, ε, του τύπου κινδυνεύουν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να κάτσουν στο δύο τραπέζι τα κόμματα επιτέλους, ώστε να μην εγκαταλείψουν την ευθύνα, την ελπίδα οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρενά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κατάσταση των δικαιωμάτων στον Μπαγκλαντέ είναι ανησυχητική. Οι εκθέσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων μα δείχνουν σε πόσο βαθμό ε, έχει οξυνθεί και κλιμακωθεί η κατάσταση. Είναι καθήκον των αρχών να εξασφαλίσουν την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω και εμεί έχουμε την υποχρέωση να επιβάλλουμε στι δικέ μα ευρωπαϊκέ επιχειρήσει συνθήκε εργασία ε, ορθές και σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν δραστηριοποιούνται στις, ε, στο Μπαγκλαντές ή άλλε χώρε. Μετά το Ράνα Πλάζα λοιπόν αντιδράσαμε, αλλά δεν κάναμε τίποτε συγκεκριμένο, ούτε νομοθετική πρωτοβουλία είδαμε από την Επιτροπή, ούτε από το Συμβούλιο κάποια αντίδραση που θα μπορούσε να μα επιτρέψει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις ε, αυτέ. Ούτε βέβαια και ρυθμιστική παρέμβαση σε σχέση με τι αποσημειώσει που θα έπρεπε, θα όφιλε να προσφέρουν αυτέ οι επιχειρήσει ούτε και ε, συνθήκες ε, αναγνώρισης ευθυνών είδαμε. Είναι πολλά λοιπόν τα πολιτικά σφάλματα, τα πολιτικά εγκλήματα και πρέπει να καταδείξουμε και τα οικονομικά εγκλήματα ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ Μπέλντερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κύριε Υπουργέ ότι πρέπει να είστε χριστιανοί στο Μπαγκλαντές ή να ανήκετε σε κάποια άλλη θρησκευτική μειονότητα. Εάν ανήκετε σε αυτή τη μειονότητα τότε φοβόσαστε για τη ζωή σας διότι οι επιθέσεις κατά χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων ε, αυξάνονται. Η ελευθερία της θρησκείας απειλείται στη χώρα. Ε, η ανεξιθρησκεία δέχεται πιέσεις φοβερές επίσημα δεν υπάρχει χώρος για τους ε, χριστιανούς να ασκούν τη λατρεία τους και βλέπουμε διακρίσεις ε, δεν σέβονται τις θρησκευτικές μειονότητες και τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα ρόλο σε αυτό Ηρίστον παρόδο ότι αγνοεί το καθεστώς της δραστηριότητα των σαλαφιστών και των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως είναι η Αλκάιντα εμείς ξοδεύουμε χρήματα για προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα τμήμα από τα χρήματα πηγαίνει για τις σκεφτικές μειονότητες. Ελπίζω ότι θα κινηθεί καταλήλως η Προεδρία. Κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, εγώ ανησυχώ, λέει Σκουκάν, για τις άνευ προηγουμένου βιοπραγίε κατά των μελών εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων, bloggers ε, που σάρωσαν τον Παγκλαντές πρόσφατα. Φαίνεται να μην υπάρχει τέρμα στις τραγικές ειδήσει που έρχονται από εκεί. Αυτές οι βίες επιθέσεις δεν είχαν σαν στόχο μόνο εκείνου που είχε αντίθετες απόψεις από τις επικρατούσες, αλλά παραβίασαν την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα. Πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Πρέπει να ερευνήσει τα εγκλήματα. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τη βεβαίωση ότι γίνονται σεβαστές οι ελευθερίες τους. Να λήξει η ατιμορρησία. Το κράτος του δικαίου πρέπει να αποκατασταθεί. Διαφορετικά, μια επιταγή εν λευκό για ριζοσπαστική συμπεριφορά και ακόλα στη βιοπραγία ε, υπονομεύει σταθερότητα του Μπαγκλαντές, κάτι που έχει συνέπειες για όλη την περιοχή, για όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Γκόμες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Τα λίμωνα Ζάριον. Λοιπόν, η κέρδισε το βραβείο Ζαχάροφ το 1994 μαζί με άλλους ε, που έχουν πάρει το βραβείο Ζαχάροφ καταδίκασαν αυτό το κλίμα βίας που επικρατεί στη χώρα έχει απειληθεί η ζωή του και δεν μπορεί να επιστρέψει και γίνονται συνεχώς δολοφονίες μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων, ε, bloggers, δημοσιογράφοι, ε, ΛΟΑΔ, ξένοι πολίτες, είναι θύματα της βίας. Πεθαίνουν άνθρωποι χωρίς να γίνονται σωστές έρευνες για να εντοπιστούν οι ένοχοι. Γίνονται πολλά εγκλήματα λοιπόν. Γίνονται αυθαίρετες δολοφονίες από πλευράς των δυνάμεων ασφαλείας ε, έχουμε σχέσεις με τον Μπαγκλαντές, έχουμε συμφωνία συνεργασίας με τη χώρα. Μετά το Ράνα Πλάζα, την καταστροφή που συνέβη, είναι απαραίτητο να αφήσουμε σε δεύτερη θέση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πρέπει να μηνύσουμε στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ότι αρνούνται την πραγματικότητα αν επιμένουν ότι το Ισλαμικό κράτο και η Αλκάιντα δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα του, Ενώ είναι υπεύθυνε αυτέ οι ομάδε για την βία Διακόπτουμε για δύο λεπτά. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικής φύσεως. Διακοπή δύο λεπτών. Συνεχίζουμε και έχει ένα λεπτό ο κύριος Μπασίρ. Κύριε Υπουργέ, είναι τραγικό για το λαό της χώρας, αλλά πρόσφατα είχαμε αυτούς τους βαρβαρικούς φόνους που μας παραπέμπουν στο μακρινό παρελθόν της χώρας για την αστάθεια και την βία. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε πέρα από το χέρι μα, ώστε ε, να μην ε, ανακατευτούμε γιατί πρόκειται για κυρίαρχο κράτος. Όμως πρέπει να καταδικάσουμε αυτή την βία και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον πολιτικό διάλογο. Ε, ο μόνος δρόμος να επανέλθει στο σωστό δρόμο η χώρα είναι τα βασικά κόμματα να δείξουν πυγμή για να βγάλουν από το διέξοδο τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνουμε υπόψη το πόσο κακή ήταν για τη χώρα αυτή η συμμαχία η κυβερνητική που έγινε γιατί ε, έφερε δυσπιστία προς τους θεσμούς της χώρας και τελικά αυτό έριξε νερό στο μήλο της ε, βίας όπως ακριβώς ε, βλέπουμε και θα πρέπει πάντως και η αντιπολίτευση να αποστασιοποιηθεί, να έχει πραγματικές πολιτικές και να μην αληθορίζει προς τους τρομοκράτες. Άρα θα πρέπει να γίνουν εκλογές και να υπάρξει υπηρεσία κυβέρνηση που να τις προκηρύξει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ένα λεπτό κύριε Παντσέρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κατάσταση στο Μπάνγκλα Ντες ε, σημαίνει ότι είναι σε πάρα πολύ άσχημη η υγεία, η ελευθερότητα, η ελευθερία και είναι πάρα πολύ κακό αυτό για τη χώρα. Γιατί έχουμε αυτέ τι ε, ενέργειε κατά των ακτιβιστών. Επομένω, δεν είναι δυνατόν εμεί να γυρίσουμε το κεφάλι προ την άλλη πλευρά. Κάνει πολύ λίγα η κυβέρνηση και επομένω θα πρέπει να τονίσουμε ότι αντικειμενικά υπάρχει κάποιο είδους συγκάλυψη των όσων εγκλημάτων κάνουν οι εξτρεμιστές. Θα πρέπει η Ευρώπη να πιέσει όσο χρειάζεται ούτως ώστε οι αρχές πιο αποφασιστικά να παρέμβουν εμείς δε ναι, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας προς τούτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο έχει τοποθετηθεί σχετικά. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει ο εκφοβισμός και η βία και η κατάσταση τα στολή των ανθρωπινών δικαιωμάτων και θα πρέπει να επιβάλλουμε σαν όρο στο Μαγκλαντές το θέμα των δικαιωμάτων. Κύριε Ζαχράντιλ τώρα για ένα λεπτό. Δεν παρίσταται. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιονγκέριος. Έχετε και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μπορούμε να πούμε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα βαδίζουν χέρι-χέρι με τα λοιπά δικαιώματα. Όπως ακριβώς είπαμε, πέρασαν τρία χρόνια μετά την τραγωδία του Ραναπλάζα. Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι πολύ λίγα έχουν αλλάξει παρά τα κέρδη που κάποιοι σώρευσαν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κάποιο είδου βελτιώσεις. Στη χώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να εκφοβήσουν τους εργαζόμενους ή εργοδότες να τους απειλήσουν με απόλυση μια που δεν υπάρχει νομική προστασία. Έχουμε επομένως όλα αυτά τα εργοστάσια για τα προϊόντα που εξάγει η χώρα, τα οποία δεν υπάγονται στην εργατική νομοθεσία. Τα ίδια τα ρούχα που φοράμε, ξέρετε, εκεί παράγονται. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα κοινωνικά δικαιώματα μου και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άλλοι τρει έχουν ζητήσει το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Σόγκορ πρώτο έχει ένα λεπτό, αλλά δεν είναι εδώ. Ο κύριο Μαριά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όπω αποδείχθηκε από τη συζήτηση, η κατάσταση στο μπαγκλαντές πραγματικά είναι εκρηκτική. υπάρχει μια συνεχής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι άλλες θρησκευτικές μειονότητες υφίστανται διώξεις. ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο ισλαμιστικό κίνημα το οποίο επιτίθεται σε δημοσιογράφους και σε μπλόγκερ. σε κοινωνικό επίπεδο το έχουμε ξαναπεί υπάρχει μια συνεχής παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων κυρίως στα εργοστάσια και από εκεί και πέρα δεν τηρούνται ούτε οι κανόνες ασφαλείας. είναι δεδομένο ότι το μπαγκλαντές αποτελεί σημαντικό εταίρο της ευρωπαϊκής ένωσης μια και εξάγει στην ευρώπη κυρίως προϊόντα κλωστοϊφαντουργίας. επομένως υπάρχει δυνατότητα από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης να ασκηθεί η επιρροή η πίεση ούτως ώστε να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα το κράτος δικαίου ο σεβασμός συνολικά της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Κονέτσνα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι στη κλωστοϊφαντουργία. 20 εκατομμύρια κατοίκων εξαρτώνται από τα έσοδα από αυτή την εργασία. 3,6 εκατομμύρια είναι οι εργαζόμενοι σε 23 εργοστάσια. Οι πιο χαμηλόμιστοι εργαζόμενοι του κόσμου, ούτε οι βασικές τους ανάγκες δεν καλύπτονται από το μισθό που λαμβάνουν. Εργάζονται για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεταθέσει όλο τον κίνδυνο στον εργαζόμενο, στο μισθωτό που εργάζεται υπό πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες γιατί υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων και πυρκαγιές και πολλοί άλλοι κίνδυνοι. Ελπίζω, είπατε, εκπρόσωπος η οποία διαπραγματεύεται με τον Μπαγκλαντές να δώσει έμφαση ιδιαίτερα και στο ρόλο των συνδικάτων και να κάνει ό,τι μπορεί για να θέσει ένα τέρμα στην κατάσταση αυτή. Παρακαλώ επόμενο Σόκο, Κύριο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Παγκλαντές φαίνεται να έχει ε, ξεφύγει από το δρόμο της δημοκρατίας και να προχωρά προς την ε, ανασφάλεια. Ο Πρωθυπουργός Σίκ Χασίνα φαίνεται να αποφασισμένος να καταστρέψει το BNP, το Bangladesh National Party της Αντιπολίτευσης πριν από τις προσεχείς εκλογές του 2018. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει ένα δρόμο αυταρχικό, ένα δρόμο εξάρθρωσης της αντιπολίτευσης και απαγόρευση και θέσεως εκτός νόμου των πολιτικών κομμάτων με αλλαγή νόμων. Ε, πολλές είναι και οι ισλαμιστικές, εξτρεμιστικές απειλές ε, με πολλές ε, επιθέσεις εις βάρος μειονοτήτων, ε, ακτιβιστών και ε, ανθρώπων της διανόησης. Κανείς δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα την ευθύνη. Ο Χασάνα κατηγορεί τον BNP βεβαίως, αλλά η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν ε, ε, εγείρει κανένα κόδωνα κινδύνου, κανένα συναγερμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να ασκήσει πιέσει στον Παγκλαντέ προκειμένου να επιβάλλει στην κυβέρνηση την προστασία των πολιτών, τους, των πολιτών της από τη βία. Ευχαριστώ. Το υπουργό ο Κούντερς έχει το λόγο τώρα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω εκφράζοντας και εγώ τον αποτοπιασμό μου για τη δολοφονία του ε, ιερέα του, των Χίντου εκφράζω συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους συγγενείς εκείνων που δολοφονούνται και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πω λίγα λόγια σχετικά με αυτά που είπατε. Όλοι ξέρουμε ότι το Μπαγκλαντές είναι περιπλοκότατη χώρα. Άκρος ευάλωτη. Από πλευράς περιβαλλοντικής είναι η πιο ευάλωτη χώρα στον κόσμο άκρο πυκνοκατοικημένη, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Εμπεριέχει πολλέ τυχέ. Έχει κάνει κάποια πρόοδο όσον αφορά του ε, στόχους, τους βιώσιμους στόχους της δείτε ποια είναι η κατάσταση κοινωνία των πολιτών στον Μπαγκλαντέ, ε, θα δείτε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο μέσω τη κοινωνία των πολιτών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει προδεύσει πολύ Έχουμε μείωση στη φτώχεια. Η θνησιμότητα των μητέρων έχει μειωθεί κατά 40% σε 9 χρόνια. Θετικά αυτά. Ταυτόχρονα εξετάζονται αρνητικότατες εξελίξεις. Συζητούνται και στο Συμβούλιο αυτές. Μειώνεται ο χώρος για δημοκρατική αντιπολίτευση και κοσμική αντιπολίτευση. Έχει πολλαπλασιαστεί η συχνότητα τρομοκρατικών επιθέσεων κατά τα μπλόγκερ θρησκευτικών μειονοτήτων και κατά των χριστιανών, αλλοδαπών, αστυνομικών, φρικτές δολοφονίες φοιτητού, καθηγητή, ακτιβιστών των LGBT, ε, γυναίκα αστυνομικού, χριστιανός μπακάλης, βουδιστής, μοναχός, δολοφονήθηκαν έχουν αυξηθεί αυτού του είδους ε, οι βιοπραγίες και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα περιορίζονται και οι πολιτικές ελευθερίες και τα πολιτικά περιθώρια για την αντιπολίτευση και για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό μας ανησυχεί, ανησυχεί και το Συμβούλιο μαζί με σας. Προφανώς, πέρα από τις δηλώσεις μας, που γίνονται συχνά, Μπορώ να παραθέσω τι έχουμε πει το τελευταίο δίμηνο. Δεν αρκούν οι δηλώσεις βέβαια. Οι δηλώσεις αναφέρονται σε γεγονότα που αναφέρατε εδώ. Ότι χρειάζεται δικαιοσύνη να αποδοθεί. Πρέπει να αντιταχθούμε στα προβλήματα. Πρέπει να καταπολεμηθεί ο βίος εξτρεμισμός, η ριζοσπαστικοποίηση. να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας την ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει η κυβέρνηση της χώρας να δεχθεί τους κινδύνους που προέρχονται από τη ρίζοσπαστικοποίηση και τους κινδύνους που δημιουργούνται από το ISIS. Διάλογος στα πλαίσια του ΙΕ αναφέρθηκε από εσά. Αυτό είναι σημαντικότατο πράγματι. Οι αντιπροσωπείες μας θα πρέπει όχι μόνο μέσω προγραμμάτων, αλλά μέσω διμερών συναντήσεων στη Σύνοδο Κορυφή ΑΣΕΜ να πλησιάσει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ και να θέσει αυτά τα θέματα. Μιλώντα για ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι, επιδεινούται η κατάσταση. Σταθερά. Ει βάρο των πλέον ευαλώτων τομέων τη κοινωνία του Μπαγκλαντέ. Πρέπει να διαβάσουμε την έκκλησή σας διότι οι δυνάμεις της τάξης κινούνται αργά και σε βιασμούς όπως σε βιασμό και δολοφονία μιας φοιτήτριας 19 ετών στην Κομίγια που ελέγχεται στατικά είναι ένα γεγονός που παραμένει ανεξήγητο. Είναι ένα παράδειγμα του πώς δεν αρκούν οι προσπάθειες των δυνάμεων της τάξης. Είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση των Μπαγκλαντές λοιπόν είναι και το σύμφωνο της βιωσιμότητας που ε, αφορά και τον Μπαγκλαντές και τις άλλες χώρες. Και αυτό τίθεται σαν θέμα. Πρέπει να συζητήσουμε ευρέω τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται με τα κοινωνικά, τα οικονομικά δικαιώματα. Μετά την κατάρρευση του Ράνα Πλάζα, όπου συνεκλώνησε τους πάντες, εδώ και τρία χρόνια, πάνω από 1.100 άνθρωποι πέθαναν, χιλιάδες τραυματίστηκαν το σύμφωνο βιωσιμότητα ήταν ε, συνήθι μεταξύ ΙΠΑ, ΑΕΛΟ, Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Μπαγκλαντέ. Εμπεριείχε τρει βασικού πυλώνε για την κλωστή φαντουργία. Είναι ένα σύμφωνο που δεν πρέπει να παραμείνει επί χάρτου, πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει και οι επιχειρήσεις να λάβουν τις ευθύνες τους για να δουλέψει το σύμφωνο, να δώσει καρπούς Χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Σεβασμό των ε, δικαιωμάτων εργαζομένων, ε, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και των συλλογικών συμβάσεων. Σημαντικό ο ρόλο συνδικάτων. Θα πρέπει να εξετάζεται η κεραιότητα των κτηρίων και η κατάσταση αφορά την υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασία και διμερώ πρέπει να το θέτουμε και στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, στι επαφέ με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ και με άλλου, να το θέτουμε υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Σημαντικότατη το Ταμείο των Δωρητών για τα έτοιμα κλωστιφαντουργικά προϊόντα και το σχετικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια δολάρια, σημαντικό ποσό που διατίθεται από το Ταμείο. Ο Καναδάς επίσης συμμετέχει τώρα πλέον σαν εταίρος. Έχει επιτελεστεί πρόοδος από τον Μπαγκλαντές. Αλλά, όπως σωστά αναφέρθηκε, υπάρχει ανάγκη η κυβέρνηση να διευκολύνει την καταχώρηση των συνδικάτων, χρειάζεται στελέχωση τη αρμόδια υπηρεσία κυβερνητική και θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να μπορεί να εφαρμόζεται και στι ε, περιοχέ εξαγωγών, με, μεταποιήσεω για εξαγωγέ. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσαι και οι συλλογικέ συμβάσει πρέπει να ισχύουν και εκεί. Είναι σημαντικό να το κάνουμε μέσω των εργαλείων που διαθέτουμε. Πρώτα απ' όλα μέσω διαλόγου που έχουμε με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ. Πρέπει να εστιαστούμε σε αυτού του τομεί, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την πρόοδο σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι ανησυχούμε για την επιδείνωση όσον αφορά τις δυνατότητες να κινείται αντιπολίτευση και ότι μειώνεται η ασφάλεια στη χώρα και θα πρέπει όλοι οι φορείς να υπομιστούν τις ευθύνες τους και η κυβέρνηση αλλά και άλλοι φορείς να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ούτως ώστε να μην συνεχιστεί η επιδείνωση της πολιτικής καταστάσεως και μέσω της βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχουμε αναπτυξιακή βοήθεια που δίδεται μέχρι 690 εκατομμύρια ευρώ χορηγείται θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματά μας ε, είναι επικαιροποιημένα όσον αφορά την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως και των εξελίξεων. Μια ερώτηση για κυρώσεις ετέθη. Δεν είμαι και φανατικός φίλος των κυρώσεων, κυρίως κατά του Μπαγκλαντές, μιλώντας βέβαια και εκ μέρους της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα λέω αυτά, έχουμε τρεις διεξόδους, τρεις δράσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε όσον αφορά τις συμφωνίες που έχουμε, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτικό διάλογο και τις ε, ελεύθερες ζώνες μεταπίσεως για εξαγωγές που είπαμε. Λοιπόν, θα είναι καλύτερο να πετύχουμε τους στόχους μας μέσω αυτών των συζητήσεων παρά να αναστείλουμε τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται για το εμπόριο. Δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε πολλά όσον αφορά τη βελτίωση της καταστάσεως για την ασφάλεια, τα πολιτικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ κύριο Κέντες, κύριε Υπουργέ. Θα παραμείνετε μαζί μας και για την επόμενη συζήτηση.